Η ημερήσια διαταξή προβλέπει την έκθεση της κυρίας ε, Γκέριγκεντ Ότεγκερ για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα έχουμε την έκθεση στην τελική της μορφή για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2014. Ε, εργάστηκα στην Επιτροπή αυτή και εργάζομαι σε αυτήν από το 2004 Οπότε παρακολουθώ πολύ προσεκτικά πώς λειτουργεί και ποια είναι τα αποτελέσματα της δράσης της Επιτροπής στην εκπόνηση νομοθεσίας. Το πώς γίνονται αντιληπτές οι αναφορές είναι μια δοκιμή για το πώς θα λειτουργήσει και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα τεράστιο αριθμό αναφορών, λαμβάνουμε συνεχώς όλο και περισσότερες, γιατί προφανώς υπάρχουν προβλήματα με την υλοποίηση της νομοθεσίας. Πρόεδρος, με συγχωρείτε. Εάν μπορείτε να πάυσετε τις παράλληλες συζητήσεις στην αίθουσα. Έχω τέσσερα λεπτά και θα ήθελα να τα αξιοποιήσω. Ο αριθμός αναφορών που λάβαμε κατά τα άλλα δείχνει ότι οι πολίτες όλο και περισσότερο έχουν συνέστηση του γεγονότο ότι μπορούν να διαμαρτυρηθούν και να προασπιστούν τα συμφέροντά του στο ευρωπαϊκό ε, επίπεδο. Το 2014 με μια διετή τάση αύξηση του αριθμού αναφορών που λαμβάνουμε, το 2014 λοιπόν είχαμε μια ελαφρά πτώση στον αριθμό αναφορών που λάβαμε στο σύνολο του έτους. Οι στατιστικές μας δείχνουν ότι το 2014 είχαμε 2.714 αναφορές, 6% λιγότερο από ότι το 2013 δηλαδή. Το 2014 περατώσαμε την εξέταση χιλίων περίπου 800 αναφορών αύξηση σε σχέση με το 2013, όμως πρέπει να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε οι αναφορές να εξετάζονται μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να δίνεται και μια ε, εύλογη λύση. Ελπίζω να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογίες πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ταχύτερα τα προβλήματα των πολιτών. Το νέο πόρταλ στο διαδίκτυο για τις αναφορές που ξεκίνησε το 2014 έκανε το σύστημα να λειτουργεί καλύτερα. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν επιγραμμικά τις αναφορές τους και ε, να συμπληρώνουν όλες τις πρωτοβουλίες που ε, τις πληροφορίες μάλλον που αφορούν το κοινοβούλιο. Επίσης λαμβάνουν ειδοποίησεις μέσω ηλεκτρονικής ε, αλληλογραφίας για οποιαδήποτε ελλαγή στην κατάσταση της αναφοράς. 80% των αναφορών που περιλήφθησαν το 2014 είχαν αποσταλεί με email και το 2014 είχαμε μια ελαφρά πτώση σε σχέση με το 13 5%. Ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που βοήθησαν στην εκπόνηση της έκθεσης αυτής και χάρη στη δική σας την συμμετοχή μπορέσαμε να έχουμε μια έκθεση πιο λεπτομερή, πιο ενδελεχή, που να αντικατοπτρίζει τη δράση τη Επιτροπή μα. Θα είμαστε διαθέσιμοι για ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο λόγο στον κύριο Αβραμόπουλο, εξωτερικό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν γέννη χαιρετίζει την έκθεση της κυρίας ε, Γκέριγκερ που ε, αφορούν τις αστιδιότητες, αφορά τις αστιδιότητες Επιτροπής Αναφορών. Από τις 790 παραδεκτές ε, αναφορές, οι 688 διαβιβάστηκαν ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, θεωρούμε ότι πράγματι, όπως λέει και η νομοδότηση, υπάρχει μια πολύ καλή ε, σχέση μεταξύ ε, των δύο θεσμών. Χαιρετίζουμε τις νέες προτεραιότητες της Επιτροπής και το πώς ορίζεται ποιο είναι ο καταλληλότερος φορέας να ανταποκρίνεται σε διάφορες αναφορές. Δεν συμφωνούμε όμως με κάποιε επιφυλάξει που εκφράζονται στην έκθεση ότι η Κομισιόν έχει επιβάλει υποτιθέμενε περιορισμούς επιτόπου σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση της ουσίας κάποιων αναφορών ή ότι πρότεινε κλείσιμο κάποιων φακέλων χωρί να αναμένει την έκβαση τη εξέταση των ζητημάτων που ετίθεντο πρέπει να σας καθησυχάσουμε και να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της και προσπαθεί να βοηθήσει ώστε να τον περισσότερο την Επιτροπή Αναφορών. Δεν υπήρξαν ποτέ επιβολές οποιοδήποτε διαδικαστικού περιορισμού. Ωστόσο, ενδέχεται να έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούσε να δώσει αναλυτική απάντηση στην ε, Επιτροπή Αναφορών, διότι δεν είχε αρμοδιότητα. Σε τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις, ε, τι κάνουμε, ενημερώνουμε την Επιτροπή Αναφορών, όπως ε, προσήκει, και οποιαδήποτε διαδικασία κλεισίματος αναφοράς ε, εναπόκειται να αποφασιστεί από την ίδια την Επιτροπή Αναφορών. Η έκθεση ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπροσωπείται στις συζητήσεις της Επιτροπής Αναφορών από, από αξιωματούχο ε, υψηλό βαθμό. Θα θέλαμε λοιπόν να σας διαβεβαιώσουμε ότι πάντοτε αποστέλουμε τους πλέον ικανούς υπά τα ζητήματα που ε, συζητούνται στην Επιτροπή Αναφορών και δεν έχουμε μέχρι στιγμής ε, λάβει ε, κάποιο σχόλιο είτε από τη γραμματεία είτε από τη, τα μέλη ότι δεν εκπροσωπήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το δέοντα τρόπο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αιτήματα για μεταφορά της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στο Εθνικό Δίκαιο. Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε προσπαθεί να διορθώσει ε, με την πιλωτική διαδικασία και τη διαδικασία επιπαραβάση ε, τις εικαζόμενες μεταφορές ε, νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τη βελτίωση θεματολογίου, έχουμε προληπτική δράση, στηρίζουμε τα κράτη-μέλη ε, στη διαδικασία εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, της ανοσιακής νομοθεσίας. Τώρα, στρέφομαι στην άμεση σχέση, ε, μάλλον στη διάθεση όλων των σχετικών εγγράφων και πληροφοριών. Θέλω να σα πω ότι πληροφορίε ό,τι αφορά χάρη διαδικασία παραβάση διατίθενται ήδη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει σε ό,τι αφορά το έργο τη στην ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση τη εφαρμογή τη νομοθεσία της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί εξηγεί το πώ ε, χειρίζεται διάφορε υποθέσει ω θεματοφύλακα ε, των Ευρωπαϊκών Συνθήκων, δηλαδή τι ε, συνέχεια δίνεται στι αναφορέ που τι διαβιβάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πληροφορίε που αφορούν τι διαδικασίε επιπαραβάση, επιπαραβάση, τι κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο δυνάμει τη Συμφωνία Πλαισίου και αποκαλύπτει πληροφορίε για διαδικασίε επιπαραβάση και στο πλαίσιο ανακοινώσεων τύπου σε ό,τι αφορά ιδίω τι αιτιολογημένε γνώμε και τι ε, παραπομπέ στο δικαστήριο. Επιπροσθέτω, ε, μπορεί κανείς να διαβουλευθεί τα σχετικά έγγραφα στην ε, βάση δεδομένων της Κομισιόν που διατίθεται στη δικτυακή πύλη. Αναζητούμε βέβαια τρόπους να βελτιώσουμε την ιχνηλασιμότητα των φακέλων. που στέλνουν ε, οι αρμόδιοι στο Κομισιόν. Έχουμε και το άρθρο 51 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι, ότι τηρείται η νομολογία του δικαστηρίου. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τις παρατηρήσεις για τις πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών, παραμένουμε δεσμευμένοι στην παρακολούθηση του έργου ε, των Ευρωπαϊκών ε, Πρωτοβουλειών Πολιτών για να επιτύχουν τους στόχους τους. Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε όπως μέχρι τώρα τα σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας αυτού του μέσου στο πλαίσιο του ισχύοντος, ε, ε της ισχύουσας διαδικασίας και πλαισίου. Σε συνεργασία με τα κοινοβούλια τα κράτη-μέλη, άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παράσχει λεπτομερέστερες πληροφορίες ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τις πτυχές αυτές ε, στην Ολομέλεια της 26 ε, Οκτωβρίου του 2015 συγκεκριμένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι θα μπορούσε ενδεχομένω να λάβει και άλλες δράσεις που θα υλοποιούνταν σε διάφορους τομείς όπως υπογραμμίζεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Όμως, τρία χρόνια μόνο έχουν παρέλθει από την έναρξη του σχετικού κανονισμού. Άρα είναι αρκετά νωρί ακόμη για να ξεκινήσει η διαδικασία νομοθετικής αναθεώρησης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει και το 2016 το έργο της για να αξιολογήσει την ενδεχόμενη ανάγκη μιας τέτοιας αναθεώρησης ή επανεξέτασης σε μεταγενέστερο στάδιο. Τώρα, ζητείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει τη συστάση του διαμεσολαβητή και να λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, ΠΕΤΗ, της Επιτροπής Αναφορών δηλαδή, για τις ε, διαπραγματεύσεις της συμφωνίας TTIP. Θέλουμε τη μέγιστη διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου αυτό μπορεί να γίνει. Χωρί βέβαια να υπονομευθεί ε, ο πυρήνα, δηλαδή η εμπιστευτικότητα, το απόρριτο που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων. Πολλές τώρα από τις συστάσεις ε, του διαμεσολαβητή, της διαμεσολαβητής στην προκειμένη περίπτωση έχουν εφαρμοστεί ή είναι στη διαδικασία. Εξετάζουμε την πρωτοβουλία πολιτών για την συμφωνία TTIP στο πλαίσιο του άρθρου 11 της Συνδίκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως δεν κατεγράφει διότι υπήρχαν κάποιοι προϋποθέσεις ε, παραδείγματο χάρη ε, σε σχέση με τον κανονισμό 211 του 2011, οι οποίε δεν τηρούνται στην προκειμένη περίπτωση. Αντιλαμβανόμαστε επίση και επαναλαμβάνουμε τη σημασία του Ευρωπαϊκού Έτου Πολιτών και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε πληροφορίε και να συμμετέχουμε σταθερά ε, στι ε, διαδικασίε τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και στο μέλλον και μέσω του διαλόγου πολιτών που διεξάγεται σε επίπεδο κρατών μελών. Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει και ε, αξιοποιεί ε, το σχετικό πρόγραμμα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης διευκολύνουμε την ε, συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών και στην Ευρωπαϊκή Διαδικασία Λήψεως Αποφάσεων. Τέλος, η Κομισιόν Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποστήριξη που έδειξε σε σχέση με το Solvit. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το Solvit θα πρέπει να τύχει περαιτέρω ανάπτυξη και συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για να αναπτυχθεί το Solvit στην πλήρη δυνατότητά του. Εν κατακλείδη. Θέλω να, να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο για την απόλυτη δέσμευση της Κομισιόν να συνεργαστεί μαζί με το Κοινοβούλιο για τα θέματα των αναφορών. Είναι ως λήθος της έννοιας του Ευρωπαίου πολίτη και βασικό δικαίωμα βασιστός ειδικών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί κύριοι βουλευτές για την προσοχή σας. Θα ξεκινήσουμε με τις πολιτικές ομάδες. Μπέκερ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών είναι ιδιαίτερα <clears throat> θετική σε σχέση με το επιτυχές έργο της Επιτροπής Αναφορών. Θα ήθελα καταρχήν να θέσω κάποια ερωτήματα σε σχέση με την έκθεση αυτή. Η λεγόμενη μεταρρύθμιση Βέλε που έγινε από το Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εξασφαλίσει μια ταχεία απάντηση και διαφάνεια. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Επιτροπής αυτής για τους εισηγητές θα εξασφαλιστεί. Θα έπρεπε να είναι σαφής η αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα έπρεπε ο ρόλος της Κομισιόν ως θεματοφύλακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπογραμμιστεί και θα έπρεπε επίσης να τονιστεί ότι η οι μετακινήσεις για έρευνα στοιχείων πολλές φορές παροχετεύονται σε πολιτική προπαγάνδα. Όλα αυτά νομίζω ότι με οδηγούν να πιστέψω ότι δεν είναι κατανοητό ότι η συγγήτρια δεν έδειξε πνεύμα συνεργασίας, ποτέ δεν ήλθε σε επαφή με μένα ως σκιώδη συγγητή και συντονιστή από την ομάδα του ΕΛΚ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγγήτρια για το γεγονός ότι δεν εμπόδισε στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων να επιτύχουν καλύτερη συνεργασία για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια λογική ψηφοφορία σήμερα. Πιστεύω ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε τον σεβασμό των συμφερόντων όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητώ λοιπόν από όλους τους βουλευτές να πούν ναι στο ψήφισμα αυτό και να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για την προάσπιση των δικαιωμάτων της. Η, η, η συγγήτρια είχε καταφέρει να αποσπάσει κάποια ομοφωνία σε σχέση με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει κυρία Καμπεθόν Ρουίς. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα της δημοκρατίας είναι η συμμετοχή των πολιτών. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή Αναφορών είναι ένα βασικό εργαλείο για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτή τη συμμετοχή και αυτό το δικαίωμα όπως ελέγχθη εδώ. Είναι πάρα πολλές οι αναφορές που έγιναν δεκτές <clears throat> το 2014 και η Κομισιόν έχει τονίσει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των πολιτών στα κράτη-μέλη και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειάζεται μια σωστή απάντηση σε όλα αυτά, αλλά φυσικά με τη σωστή διαδικασία και εγκαίρος. Επομένως θα πρέπει να συμμετάσχει όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φυσικά και η Κομισιόν και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών για να υπάρξει ένα σαφές μήνυμα ότι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο, στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσει σε μια ανακοίνωση που καθορίζει σαφώς τις υποχρεώσεις κάθε μία από αυτές τις εμπλεκόμενες πλευρές στη διαδικασία αναφορών. Ευχαριστώ ο κύριος ε, Μαριά από το ΙΣΙΑ. Πρόεδρε, η Επιτροπή Αναφορών αποτελεί το θεσμικό όργανο στο οποίο οι πολίτε τη Ένωση μπορούν να προσφύγουν για την προάσπιση των δικαιωμάτων του και τον έλεγχο τη σωστή εφαρμογή του δικαίου τη Ένωση. Η Επιτροπή Αναφορών έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα φόρουμ διαλόγου ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα εξουσίας της Ένωσης και των κρατών μελών τη και τους ίδιους τους πολίτες. Μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της Επιτροπής Αναφορών είναι αυτή του Οκτωβρίου 2015 η οποία έκανε αποδεκτή την εισήγησή μου να κριθεί παραδεκτή η αναφορά των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης πααe για το ζήτημα των οφειλών της γερμανίας προς την ελλάδα. έτσι καλείται πλέον για πρώτη φορά η γερμανία να τοποθετηθεί δημόσια σε ένα ευρωπαϊκό δικαιοδοτικο όργανο όπως είναι η επιτροπή αναφορών για το ζήτημα των πολεμικών επαναρθώσεων του αναγκαστικού κατοχικού δανείου των αποζημιώσεων των συγγενών των χιλιάδων ελλήνων πολιτών που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και αυτών που δολοφονήθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αρχίζω την παρέμβαση τονίζοντα ε, τη μεγάλη σημασία τη επιτροπή Αναφορών για τη συμμετοχή Δημοκρατία και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια θηρίδα ανοιχτή για του πολίτε. Πάνω από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουμε μεταξύ μα κάποιου από αυτού, έρχονται, μπορούν να ε, υποβάλουν απευθεία στα αιτήματά του. και αυτό έχει μοναδική αξία. Υπάρχουν κάποιε ε, ανησυχίε ότι αφορά τη δικαιοσύνη, το περιβάλλον, δική αγορά, θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτά είναι τα, τα αντικείμενα των περισσότερων αναφόρων. Πρέπει να το έχουμε υπόψη. Χώρε όπω η Ισπανία. Είναι ανησυχητικό που σε ό,τι αφορά τον αριθμό αναφόρων εξακολουθούν να είναι στην κορυφή και βέβαια σε ό,τι αφορά τον αριθμό παραβάσεων. Μεταξύ αυτών είναι και η Ελλάδα και η ε, Ιταλία, οι χώρε από τι περισσότερε παραβάσει. Θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμό και συνεργασία τη Κομισιόν με άλλα όργανα και θεσμού τη Ένωση, αλλά και με τα εθνικά κοινοβούλια και τι επιτροπέ τη κοινοβουλευτική Βασική πρόκληση είναι να έρθουμε στο ύψο των προσδοκιών των πολιτών και να είμαστε αποτελεσματικοί για να προσπίσουμε τα δικαιώματά του. Ε, η παράγραφο 21 είναι σημαντική. Λέμε ότι ο χάρτη των δικαιωμάτων λυπόμαστε που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί από όλα τα κράτη. Υπάρχει ε, σύγχυση ό,τι αφορά την εφαρμογή του χάρτη. Η αυστηρή ερμηνεία του άρθρου 51 του χάρτη, ε, του οποίου πολλές φορές δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ότι δεν μπορεί να δράσει στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πρόκληση και με κοινή προσπάθεια θα πρέπει να υπερπηδήσουμε τα σχετικά εμπόδια στο συνάδελφο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν πάρα πολύ γρήγοροι, λέει η πρόεδρος. Γκουσμάν και σας παρακαλώ να μην μιλάτε τόσο γρήγορα οι υπόλοιποι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε με την πλάτη προ του πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση, σκεφτόμενη μόνο το συμφέρον του χρηματιστηριακού κεφαλαίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Κοινοβούλιο όμω και αυτό είναι πολύ μακριά από του πολίτε μα. <clears throat> Οι ευρωπαϊκοί δεσμοί δεν είναι δημοκρατικοί και δεν αντιμετωπίζουν πραγματικέ ανάγκε των Ευρωπαίων. Και αυτό είναι πραγματικότητα όταν δούμε ποιε είναι οι πολιτικέ οι οποίε επιβάλλονται που υποστηρίζουν την οικονομική ελίτ και μόνο. Γι' αυτό ο μόνος τρόπος να υπάρξει επαφή αυτών των θεσμών με τους πολίτες είναι η Επιτροπή Αναφορών. Μόνο μέσω των αναφορών που παρουσιάζονται που μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα πόσο μεγάλη είναι η απόσταση η οποία υπάρχει μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της πραγματικότητας. Είμαστε έτη φωτός από τους ανθρώπους που υποτίθεται εκπροσωπούμε. Δεκάδες αναφορές ουσιαστικά ε, έχουν τονίσει ότι πρέπει να απορριφθούν τα διαιτητικά δικαστήρια που επιτρέπουν στις ε, πολυεθνικές εταιρείες να αγνοούν τα εθνικά δικαστήρια. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κοφεύει και ζητεί να συνεργαστούν οι διαπραγματεύσεις για αυτές τις συστήκες που έχουν γίνει, έχουν εραφτεί στα μέτρα των μεγάλων πολυεθνικών. Οι αναφορές επίσης ζητούν να σταματήσει μια πολιτική για τη μετανάστευση που αντιβαίνει στην πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά η Ευρώπη εξακολουθεί να ασκεί τη βία, τις ε, απελάσεις και τα κλειστά σύνορα. Επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των Ευρωπαίων και η μόνη συμμαχή της είναι τα άλλη. Τέρμα ο χρόνος σας κυρία Βουλευτής, λυπάμαι πάρα πολύ. Μιλάτε και πολύ γρήγορα εξάλλου. Ρέντα δύο λεπτά από τους πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και του συναδέλφου για την εξαιρετική δουλειά στην έκθεση αυτή, με τη συναντήση των σκιωδών από όλε τι ομάδε, να μπορούν να κάνουν τη φωνή του να ακουστεί. Ε, είναι ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα το οποίο δεν αμφισβητείται εδώ, διότι η δράση τη Επιτροπή των Αναφορών γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Η μεταχείριση των αναφορών μπορεί να διαμορφώσει την στάση προ την Ευρωπαϊκή Ένωση για πάντα από την πλευρά των πολιτών. Και είναι πολύ σημαντικό πώ απαντάμε στου πολίτε, όχι όμω ει βάρο τη ποιότητα τη δουλειά μα. Πρέπει επιτέλου να δούμε το πόσο μεγάλο φόρτο εργασία έχουμε με τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών και να αξιοποιήσουμε του πόρου που διατίθενται σε αυτή την Επιτροπή. Πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία αναφορών έχοντα υπόψη τα συμφέροντα του αναφέροντο. Δηλαδή να είναι σαφεί και ξεκάθαροι κανόνε για την παραδεκτότητα των αναφορών. Έχουμε καταβάλει πρόοδο ω προ την ε, τα κατεύθυνση αυτή με το πόρταλ για τι αναφορέ, αλλά ακόμη υπάρχουν ελλείψει και κενά που πρέπει να καλυπτούν για να έχει το, η πύλη αυτή στο διαδίκτυο μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για του πολίτε Πρέπει επίση να παρακολουθήσουμε τι εξελίξει να δούμε πώ συμμετέχουν οι υπόλοιπε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ στην δράση των αναφο... Αναφορών όταν ε, το μισαρμοδιότητα είναι κοινή και να ληφθεί πιο σοβαρά υπόψη η Επιτροπή αυτή ω ε, θεματοφύλακα των συνθήκων. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έπρεπε να επαναλαμβάνει ότι λένε οι αρχέ των κρατών μελών, διότι ω θεμελιώδη δικαίωμα η αναφορά πρέπει και ω τέτοιο να αντιμετωπίζεται. Δυστυχώ, κάποιε φορέ η έλλειψη πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι που αντικατοπτρίζεται και στην άλλη περίπτωση τη πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, η αφοσίωση λοιπόν θα κρυθεί από το κατά πόσον τα εργαλεία που προβλέπουμε για τη συμμετοχή των πολιτών δεν δεν παρακολύονται από τεράστιους φραγμούς που προβλέπονται για την πρόσβαση. Έχει επικριθεί και από τον Ευρωπαϊκό Δημοσιολαβητή η τάση αυτή και τον ευχαριστώ για την, ε, με την ευκαιρία αυτή γιατί ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, έχει περισσότερη λογοδοσία και να συνεργάζεται περισσότερο με του πολίτε. Τα συμφέροντα των πολιτών λοιπόν πρέπει να καθοδηγούν στο έργο του την Επιτροπή των Αναφορών, το Κοινοβούλιο και όλα τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό η κυρία Εύη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να ξεκινήσω από ένα άλλο δεδομένο, το δεδομένο των παραδεκτών αναφορών που είναι το 39% των αναφορών που λαμβάνουμε συνήθως. Προφανώς ε, το στοιχείο αυτό δείχνει ότι δεν κατανοούμε πλήρως και ότι υπάρχει σύγχυση για το ποια είναι τα πεδία δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, ε, πρέπει να μάθουν πολύ καλά όλοι οι πολίτες ποια είναι τα δικαιώματά τους ε, στην αναφορά. Θα έπρεπε όλοι να μπορούν να το αξιοποιήσουν. Άρα ο βασικός στόχος είναι να επιληθούν τα διάφορα προβλήματα που εντοπίζουν οι πολίτες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και εμείς από την οπτική γωνία των ε, κοινοτικών οργάνων θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δώσουμε αποτελεσματικές απαντήσεις. Να τονίσω και εγώ πως ε, η πύλη στο διαδίκτυο ακόμη και σήμερα δεν λειτουργεί επαρκώς. παρόλα αυτά είναι ένα σημαντικό εργαλείο που ε, έχει προβλεφθεί και για την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών που τελικά όμως αποδείχθηκε μια εξαπάτησή τους. Ευχαριστούμε. Γκόντιν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η δράση της Επιτροπής Αναφορών έχει επιβραδυνθεί το 2014 με 2.714 αναφορές. Μια πτώση κατά 6% σε σχέση με το 2013. Βλέπουμε ότι πρέπει με τις επιπλέον αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή Αναφορών να προβλεφθούν και τα απαραίτητα μέσα. Το 2014 οι 1070 αναφορές κρίθηκαν μη παραδεκτές, 817 παραδεκτές και πολύ λιγότερες ε, περατώθηκαν. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι το δικαίωμα στην αναφορά για επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πολύ γνωστό στους πολίτες. Θα πρέπει να δούμε και την πολιτική διάσταση του θέματος πέραν της νομικής και τεχνικής και θα πρέπει να κοιτάξουμε να ε, προβλέψουμε για τους πολίτες τη δυνατότητα προάσπισης των συμφερόντων τους. Η συμμετοχική δημοκρατία με τις πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών είναι κάτι που θέλουμε να προαχθεί, αλλά βλέπουμε το συγκεκριμένο εγχείρημα της πρωτοβουλία να αποτυγχάνει. Δεν ε, μπορούν να ανακληθούν ε, ή να καταργηθούν νομοθετικά κείμενα, ούτε να πάψει το, ε, η προπαρασκευαστική φάση τη εκπόνηση νομοθεσία. Οπότε η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών καθίσταται κενή νοήματο ακόμη και με τις διαμαρτυρίες για το TTIP και παρά τα 3 εκατομμύρια υπογραφές που συλλέξαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να δεχθεί την πρωτοβουλία αυτή ε, λέγοντα ότι οι διαπραγματεύσει για τη συνθήκη δεν είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, και όμω υπάρχει ένα προηγούμενο, διότι το 2013 με την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποδεχθεί την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα επιχειρήματα που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολιτικού χαρακτήρα. Όταν καταγράφει τέτοιε πρωτοβουλίε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τίποτε δεν γίνεται. Το είδαμε με τα πειράματα σε ζώα ή το δικαίωμα στην υδροδότηση. Οι Ευρωπαϊκοί πολίτε έτσι αποθαρρύνονται και στρέφουν τα νότα στι ε, δικασίε όπω η το δικαιωμα στην υδροδοτηση οι ευρωπαιοι πολιτε ετσι αποθαρρυνονται και στρεφουν τα νοτα στι δικασιε οπω η πρωτοβουλίε των Ευρωπαίων Πολιτών και η Επιτροπή Αναφορών. Η έκθεση ε, Γκέτιγκερ πολύ σωστά εντοπίζει τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστούμε κυρία Μουρβάη για 1,5 λεπτό. Η έκθεση αυτή για το έργο της Επιτροπής Αναφορών δεν έχει καμία σχέση με τη δική μου προσωπική εμπειρία στρέφομαι γι' αυτό λοιπόν ε, στον, προ, ε, στον παρόντα επίτροπο ε, και θέλω να τον παρακαλέσω να εξηγήσει. Δεν φοράει τα ακουστικά του βέβαια, φαίνεται να καταλαβαίνει τέλεια τα ουγγρικά. με ακούει λοιπόν πολύ προσεκτικά, γιατί και γι' αυτό το, το, το λόγο άλλωστε βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, θα ήθελα Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, να σας δώσω όταν έρθω στο βήμα ένα έγγραφο σε Α4. Ουσιαστικά πρόκειται για αντίτυπο μιας απόφασης της Επιτροπής Αναφορών ε, για τα ε, θύματα στεγαστικών δανείων ε, πολιτών συγκεκριμένα, δάνεια σε ξένο νόμισμα. Πρόκειται για εκατοντάδες πολίτες που εξαπατήθηκαν από τράπεζες για να συνάψουν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο ή άλλα νομίσματα υπεγράφουν οι αναφέροντες ε, μια δεκαπεντασέλιδη αναφορά ε, συνταγμένη από δικηγόρους και έχουν λάβει και μια απόφαση, ε, μια απάντηση συγγνώμη, η οποία όμως δεν ξεπερνάει τη μισή σελίδα. Όταν λέτε λοιπόν ότι κάθε αναφορά εξετάζεται με διαφανή τρόπο και ως μοναδική περίπτωση. Πώς αυτό συνάδει με τη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή ε, σε μια τόσο μακροσκελή πολυσέλιδη αναφορά να πάρουν απάντηση μισή σελίδα σε αναφέροντες Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Γιάρ. Θετική είναι εν γέννη ε, η δράση Επιτροπή Αρβόρ. Θα ήθελα όμω να τονίσω τρει ε, πτυχέ σε σχέση με αυτό που και ο κύριο ε, Μπέκερ μόλι πριν. Πρώτα απ' όλο πολύ σημαντικό να αποφασίσουμε γρήγορα για παραδεκτές και μη παραδεκτές αναφορές για τι οποίε δηλαδή, δεν έχουμε εμεί αρμοδιότητα και τις οποίες δεν θα πρέπει να εξετάσουμε γιατί αυτό θα συνιστούσε δαπάνη χρόνου ενώ έχουμε αρμοδιότητα για άλλες αναφορές και θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με αυτές. Δεύτερον, θα πρέπει να τηρούνται οι προθεσμίες. Αυτό είναι κάτι ε, το οποίο ε, προβλέπεται και με τη μεταρρύθμιση ΒΕΛΕ. Εννέα μήνες αφού το επιλαμβάνεται ε, της η, η Επιτροπή Αναφορών πρέπει να έχει γίνει πρώτη συζήτηση, να έχει ληφθεί πρώτη απόφαση. Επίσης, κατά τρίτον, υπάρχουν ε, κάποιες περιπτώσεις όπου οι βουλευτές, τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών θεωρούν ότι θα πρέπει να βελτιωθεί νομοθεσία. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με άλλες επιτροπές και πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία αυτή. Όχι όμως μόνο αυτό και η συνεργασία μεταξύ της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου και άλλων Εθνικών Κοινοβουλίων. Θέλω να ευχαριστήσω ε, τη Γραμματεία και τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών. Δεν είναι εύκολο να είναι κανείς ε, μέλος της Επιτροπής Αναφορών πάντοτε. Η Επιτροπή Αναφορών για μένα είναι ένα δείγμα δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν έτσι οι πολίτες να αναφέρονται άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, είναι ένα είδος σεισμογράφου της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Θα πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ και στον Επίτροπο και στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν θέλουμε να ακούσουμε άμεσα τη φωνή των πολιτών αψημίθευτη και καθαρή, τότε πρέπει να διαβάσετε τις αναφορές που μας απευθύνονται. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντάρλινγκ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι θαυμάσιο το γεγονός ότι οι εκλογές μας έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για περιπτώσεις που δεν υπόκειται σε δικαστική διαδικασία που θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί. Την πρώτη μου χρονιά στην Επιτροπή Αναφορών έχω ακούσει σαφώς τη φωνή των πολιτών από όλη την Ευρώπη και ένα από τα θέματα που τους ε, απασχολείται το θέμα της τύπη παραβίας των δικαιωμάτων των πολιτών και ιστορικές περιπτώσεις για λανθασμένη απόφαση της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, όπως την περίπτωση των απεργών για τα ορχεία του Καμελέκ. Πολλές φορές όμως έχουν εμποδιστεί οι αναφορές αυτές με το να ακούμε αυτά τα οποία λένε οι πολίτε μα, <clears throat> η Επιτροπή Αναφορών έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Γι' αυτό το λόγο, εμεί θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο το ρόλο τη Δημοκρατία μέσω τη Επιτροπή Αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δώσουμε περισσότερε δυνατότητε στου βουλευτέ να ακούν την άποψη των πολιτών και να του εξυπηρετούν με τον τρόπο αυτό. Ένα λεπτό, κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία και όλου του συναδέλφου για την πολύ καλή του δουλειά και για, τη... για το πνεύμα συμβασμού που έδειξαν αυτή την εβδομάδα στην έκθεση αυτή. Η Επιτροπή των Αναφορών, ε, τη οποία είμαι πρόεδρο, είναι ε, μια γέφυρα την ε, σχέση πολιτών ευρωπαϊκών οργάνων. Θα έπρεπε να επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλουν τις ιδέες και τις παρατηρήσεις τους στους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σήμερα η έκθεση αυτή εντοπίζεται στη δράση της Επιτροπής για το 2014. Μια ειδική χρονιά, διότι ήταν ε, χρονιά εκλογών για το Κοινοβούλιο και βεβαίως αυτό επηρέασε και τη δράση της Επιτροπής μας. Με μεγάλη χαρά ε, βλέπουμε ότι εντοπίζεται το γεγονό ότι και η Γραμματεία και η διευθυντές και υπεύθυνοι τμήματάρχες της Επιτροπής Αναφορών βελτίωσαν το έργο τους το 2014. Οι μέθοδοι εσωτερικής εργασίας εξυγχρονίστηκαν από το 2014 και ήδη φέτος έχουν φέρει τους πρώτους καρπούς. Θεωρώ ότι είναι θετικό το γεγονό ότι πείσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει τον πρώτο τη ε, αντιπρόεδρο ω επίτροπο για να συνεργάζεται μαζί μα. Και θα συνεργαστούμε, ε, πιστεύω, όλοι στενά σε μνημονικό πνεύμα για να βοηθήσουμε να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των πολιτών με τη δράση μα. Ευχαριστούμε, κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την ε, συνάδελφο για την εξαιρετική έκθεση. Δεν θα επαναλάβουμε όσα υπόθηκαν ήδη, απλώς να πω ότι σήμερα έχουμε πολύ καλύτερη συνεργασία, ιδιαίτερω ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Και να ευχαριστήσω και ε, το δημοσιολαβητή για την δουλειά του ως τώρα. Χρειάζονται όμως και κάποιες βελτιώσεις. Δεν έχουμε αρκετά μέσα ούτε πόρους για να καλύψουμε τις ε, αρμοδιότητες και τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προβλεφθούν περισσότερα. Και νομίζω ότι δεν έχουμε ακόμη αρκετές μελέτες, επιτόπου μελέτες, ε, και νομίζω ότι και αυτή η διάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί. δεν έχουμε επιτροπή αναφορών ε, ε, που να είναι ε, απολύτως ανοιχτή όπως θα θέλαμε. Οι πολίτες θέλουν να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει και θα πρέπει να φροντίσουμε οι πολίτες να συμμετέχουν περισσότερο στην δουλειά μας. Κάποια από τα μέλη της Επιτροπής δεν είναι αρκετά δραστήρια. Ευχαριστούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον που βλέπουμε την αντίσταση κατά της TTIP στο έγγραφο αυτό και αυτό είναι και ενθαρρυντικό. Πολλοί από τους εκλογείς μου μου έγραψαν εκφράζοντα τις ανησυχίες τους σε ό,τι αφορά τη συμφωνία TTIP ότι θα ανοίξει την, ε, την ε, Αγγλική Υπηρεσία Υγείας σε ιδιωτική σε ιδιωτικό ανταγωνισμό και επίσης η διαδικασία διαρρύθμισης διαφορών θα πάρει την εξουσία από τα δικαστήρια και θα δώσει την εξουσία σε αυτού που επιζητούν κέρδη. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί έσχο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα καταλάβετε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι εν ώψη της TTIP ε, θα πάρουν θέση στο δημοψήφισμα για το Brexit. Αν θέλετε λοιπόν να φύγετε από, το, από την TTIP θα πρέπει να βγείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν γίνει το δημοψήφισμα. Βαλέντσα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω τη συμφωνία της ετήσιας έκθεσης για τις δραστηριότητε επιτροπής μας. Όχι μόνο να μας δίνει μια πλήρη εικόνα για το τι έχει γίνει το 2014, αλλά εκπροσωπεί επίση και ένα οδηγό για το μέλλον, για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις ε, αναφορές στο μέλλον. Είναι δικαίωμα όλων των πολιτών να καταθέτουν αναφορές. Αυτό έχει να κάνει και με την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να έχουν οι πολίτες στην, στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αναφορές είναι ένα από τα κύρια εργαλεία για τους πολίτες μας να είναι καλύτερα εμπεπλεγμένοι στη δημοκρατική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν σχετικά ότι οι τροπολογίε του ΕΛΚ είναι πάρα πολύ σημαντικές στην εκθεσία αυτή γιατί καταδεικνύουν σαφώς ποια είναι η υποχρέωση να τηρηθούν οι διοικητικές διαδικασίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πολλές φορές ξεχνάμε ότι αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ σημαντικές στο έργο μας. <clears throat> Πρόκειται για κατευθυντήριες αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν όλο το κύκλο των ε, αναφορών και να εστιάσουμε στα πραγματικά αποτελέσματα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι και να κάνουμε δεν δίνουμε φρούδες ελπίδες στους ε, αναφερόμενους. Θα πρέπει να είμαστε διαφάνει στον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζουμε και ότι τα θέματα των πολιτών πράγματι αντιμετωπίζονται στην Επιτροπή μας και θα πρέπει να μειώσουμε τη δυνατότητα να πολιτικοποιηθεί η ημερησία διάταξη της Επιτροπής Αναφορών. Αυτά είναι λοιπόν τα πρακτέα στην Επιτροπή μας. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη και να βρούμε μια σωστή ισορροπία και σωστό ορισμό <clears throat> της, ε, του αποδεκτού των αναφορών και το σωστό τρόπο για να εξηγούμε στους αναφερόμενους γιατί κάποιες φορές δεν είναι παραδεκτές οι τροπολογίες τους, οι αναφορές συγγνώμη, ή πρέπει να κλείσουν κάποτε. Κυρία Τζίφριντα, για ένα λεπτό. Η Επιτροπή Αναφορών έχει έναν θεμελιώδη ρόλο να προσεγγίζει τους πολίτες τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι το front office ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι η Επιτροπή των Αναφορών που κάνει το Κοινοβούλιο πραγματικά δημοκρατικό θεσμικό όργανο. Ξέρουμε πραγματικά πώς γίνεται αντιληπτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολύ απόμακρη συχνά. Οι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι συμμετέχουν στι όλε τι διαδικασίε μόνο κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών. Όμω η δράση τη Επιτροπή αυτή δεν εξυπηρετεί μόνο του πολίτε, αλλά είναι καθοριστική και για μα. Κοιτάζοντα τα θέματα που θίγονται από την Επιτροπή Αναφορών, καταλαβαίνουμε τι διακυβεύεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πρέπει να αλλάξει. Υπάρχουν αιτήματα στις αναφορές που πρέπει να γίνουν προτεραιότητες για μας. Αλλά είναι απαράδεκτο οι αναφορές να εξετάζονται με σημαντική καθυστέρηση, κάποιες φορές και ένα χρόνο μετά την αποστολή τους. Πρέπει να προωθεί ένας τρόπος για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα που μπορεί να καταστήσει κενό νοήματος το το, ε, την ίδια του την ουσία και τον αρχικό του στόχο. Θα πρέπει λοιπόν οι υπάλληλοι συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής που εργάζονται αδιάκοπα να υποστηριχθούν. Ευχαριστούμε κυρία Πίτερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή Αναφορών προστατεύει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών όπως τα όπως θεμελιώνονται στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Και συνήθως υποβάλλονται αναφορές ως προς το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζει τη ζωή των πολιτών. Θα έπρεπε λοιπόν να επιλύουμε τις ε, δυσχέρειες στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της δράσης της Επιτροπής αυτής. Η Επιτροπή Αναφορών διαρκώς βελτιώνει την ε, μεθοδολογία της και η ομάδα μου έχει υποβάλει μια τροπολογία ώστε να αναφερθεί ότι τα κάτι μελη θα πρέπει να κινητοποιηθούν περισσότερο για να εφαρμόζουν ε, τα όσα προβλέπονται για επιτροπές αναφορών στα δικά τους εθνικά κοινοβούλια. Αυτό συζητήθηκε πέρυσι και σε κοινή συνεδρίαση με τα μέλη τη Επιτροπής Αναφορών. Δεν έχουν βεβαίω όλες οι συνελεύσει την ίδια δομή σε όλες τις ε, χώρες. Όμω θα ήταν ιδανικό εάν υπήρχε συνεργασία τη Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τι ομόλογέ του επιτροπέ τη Εθνικέ Βουλέ. Εδώ λοιπόν θα διευκολυνόταν πάρα πολύ η δουλειά της δικής μας επιτροπή Επιτροπής Αναφορών. Όσο αφορά επίσης τη φροντίδα των παιδιών, τα παιδιά δεν τα αναλαμβάνουν μόνο γονείς που μπορεί να έχουν πάρει διαζύγιο, αλλά και κάποιε φορές άλλοι άνθρωποι που αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους. Κατά κάποιο τρόπο αυτό ισχύει και για την Επιτροπή ε, Αναφορών εφόσον ε, και αυτό το θέμα είναι κάτι που εξετάζει η Επιτροπή Αναφορών. Πρέπει λοιπόν η διαδικασία να παραμείνει ανοιχτή ώστε να μπορούμε να ε, προτείνουμε μια απόφαση για το θέμα αυτό. Εάν οι τροπολογίες ε, που εντοπίζουν τα ζητήματα αυτά δεν περάσουν, δεν θα έχει και νόημα στη λειτουργία της Επιτροπή Αναφορών. Ευχαριστούμε για τη λεπτό κύριο Τσάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να διατηρήσουμε το δικαίωμα στην αναφορά. Αυτό είναι ένα εργαλείο επικοινωνία για του πολίτε. Οι αναφορέ είναι η πύλη προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του ευρωπαϊκού θεσμού. Θα πρέπει αυτό να εξυπηρετεί του πολίτε. Στην έκθεση αυτή βλέπουμε όμω ότι σε σχέση με το σύνολο των αναφορών υπάρχουν λίγες αναφορές και η δική μου εμπειρία είναι η ίδια ως μέλος της ε, ουγγαρόφωνης μειονότητας στην Σλοβακία βλέπω να μην υπάρχουν πολλές αναφορές από τη δική μας πλευρά. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι πιο συχνά αντικείμενο αναφορών η ελευθερία διακίνηση το περιβάλλον, οι διοικητικέ τη λειτουργίε, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ενδιαφέρουν του πολίτε. Είναι οι κύριοι τομεί που θα πρέπει να αντιμετωπίζει η Επιτροπή Αναφορών. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην δημιουργία συνειδητοποίηση. Πολλοί πολίτε δεν ξέρουν τίποτα για τα δικαιώματά του. Οι στατιστικές των προηγουμένων ετών δείχνουν ότι είναι πολύ λίγε οι αναφορέ από την Ουγγαρία ή από την Σλοβακία. Ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών προσπαθώ να φέρω λοιπόν το έργο της Επιτροπής Αναφορών στο λαό της χώρας μου. Το δικαίωμα στην αναφορά είναι ένας τρόπος για να ασκηθεί έλεγχος στην διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκθεσία αυτή όμως δεν μιλάει καθόλου για τις εγγύησεις οι οποίες θα βελτίωναν το έργο της Επιτροπής Αναφορών. Η διοικητική μεταρρύθμιση η οποία εισήχθη από το Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αντανακλά αυτήν την διαδικασία. Πιστεύω όμως ότι μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία της Επιτροπής και τον σεβασμό των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Catch the eye. Ξεκινώ με την κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ε, πω ότι είναι πάρα πολύ καλή δουλειά της Επιτροπής Αναφορών. Ήμουν και εγώ ε, μέλος κατά παρελθόν ασχολούμαι με τις αρπαγές παιδιών αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά ε, σε αυτό το τομέα. Το είπε και ο προλαλής σας. Οι αναφορές που αφορούν τα παιδιά είναι πολύ δύσκολε, ιδίως όταν μιλάμε για θεσινοριακές υποθέσει και όλο και περισσότερε υποθέσει θα έρχονται ε, στην Επιτροπή μας. Θέλουμε ε, να δώσουμε κάποια καθοδήγηση στα άτομα αυτά που υποφέρουν. Και αυτές είναι ε, οι πλέον συναισθηματικά φορτισμένες και δύσκολες αναφορές. Ζητώ λοιπόν να συνεχιστεί η συνεργασία μας, ώστε το γραφείο μου, που επαλαμβάνω ασχολείται πλέον με την αρπαγή των παιδιών και η Επιτροπή Αναφορών, να συνεργαστεί και για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες 2 που είναι σημαντική σημαντικό νομικό κείμενο. κυρία Βαλίνα τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Με βάση το Μέτρο του Μαΐου 2015, η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ένωση δεν ξεπερνά το 40% και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, στην κρίση των προσφύγων, τις πολιτικές λιτότητας της Τρόικα, στην εγκατάλειψη της υπαίθρου, την υπάσπιση του φράκινγκ, της υδρορογμάτωσης, αλλά και το ότι δεν ε, στηρίζονται ε, προσπάθειες εξάλληψης νόσων όπως ε, η πατήτη γάμα και άλλες. Πρέπει να, πρέπει να κάνει πιο πολλά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δίνει πραγματικά τη δέουσα προσοχή να μην στρέφει άλλο και να δώσει πραγματικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα. Να μην είναι απλοί τεχνοκράτες ε, στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Κύριε Αβραμόπουλε, πρόεδρος, επαναρχόμαστε. Βλέπετε ότι έρχονται οι συνάδελφοί μας. Ε, θα πρέπει να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά για να γίνετε, για να Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, εκφράσω τι ευχαριστίε μου την κυρία Γκέριγκερ Ντε για την έκθεσή της. Και να ευχαριστήσω και τους βουλευτές που πήραν το λόγο σε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σημειώσαμε ιδιαίτερη προσοχή όλα τους τα σχόλια. Το δικαίωμα του αναφέρεστε είναι θεμελιώδης δικαιώμα των πολιτών βάσει των συνθήκων. Το να δείξουμε στους πολίτες ότι τις μεριμνές τους τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη είναι ένας τρόπος για να ενισχύσουμε την πίστη τους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Αναφορών για να βεβαιωθεί ότι υπάρχει δραστική και αποτελεσματική μεταχείριση των αναφορών. Ε, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ η κυρία ε- Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ως ε, κύρια εισηγητρία για το θέμα αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα για τη δυνατότητα που είχα να συγκροτήσω μια έκθεση η οποία είχε πολλές φιλοδοξίες και πολλές συμβολές από τους συναδέλφους. Νομίζω ότι καταδεικνύει την τωρινή κατάσταση της εργασίας της Επιτροπής μας και έχει και προτάσει για το μέλλον. Ο στόχος της έκθεσης είναι η περαιτέρω βελτίωση του έργου μας για τις αναφορές. Κάποιοι από εμά μπορεί να έχουν επικρίσεις σε σχέση με ορισμένες ε, ε απόψεις για την ε, έκθεση αυτή, αλλά αυτό <clears throat> είναι καλό, είναι θετικό. Δείχνει ότι υπάρχει μια πολυφωνία, δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα τομείς στους οποίους εμείς θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο και εμείς θα κάνουμε όλα αυτά τα οποία θα μας φέρουν κοντύτερα στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και ελπίζω θα οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματικό έργο της Επιτροπής Αναφορών προς όφελος των πολιτών μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για τις λεπτομερείς εξηγήσεις του και νομίζω ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών πολλών ανθρώπων. Χρησιμοποιώ λοιπόν και αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές μου γιατί ήταν πολύ χρήσιμες οι παρατηρήσεις τους Μπέκερ, Αλμπιόλ, Εύη, Μπετσέρα, Μαριάς, Ρέντα. Όλους αυτούς θέλω να ευχαριστήσω και επίσης θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συντονιστές, συμβούλους, το προσωπικό της γραμματείας που εργάστηκαν για αυτή την εργασία και τον κύριο Καμπεθόν Μπάιρ Κύρκος Λεκόκ Περές και την ε, βοηθό μου την κυρία Μπέρσχα παρά τις αρχικές ε, δυσκολίες και διαφορές μπορέσαμε να υποβάλουμε μια αξιόπιστη έκθεση για το μελλοντικό έργο της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Πέρα τη συζήτηση η ψηφοφορία θα γίνει